Ladies Κυρίες και κύριοι, κυρίες και κύριοι, αν θέλετε να βγείτε από το ημικύκλιο, παρακαλώ εξέλθετε το συντομότερο της αιθούσης, γιατί θα θέλαμε να αρχίσουμε τη σύνοδο. Uh, ladies and Κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι, σας παρακαλώ, μην κάνετε ιδιωτικές συζητήσεις στην Ολομέλεια. Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε, θα ξεκινήσουμε σε 30 δευτερόλεπτα. Παρακαλώ συνάδελφοι, επαναλαμβάνει ο Πρόεδρος, καθίστε για να μην αναγκαστείτε στο τέλος να μείνετε περισσότερο. Δώστε μας τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε με τη συνεδρίασή μας τώρα. Wznawiam Θα ήθελα να ξεκινήσω με κάποιες ανακοινώσεις. Πρώτα απ' όλα, έχουμε πληροφορίες και σταματήστε να μιλάτε όσοι εδώ κάνετε πηγαδάκια μέσα στο μικύκλιο. Άμα θέλετε να αποχωρήσετε, αποχωρήστε τώρα. Γρήγορα. Εγώ σας καλώ να καθίσετε για να συμμετάσχετε. Αλλά αν δεν θέλετε, όχι πηγαδάκια στην αίθουσα. Πολωνικά ο πρόεδρος τώρα. Δυστυχώς έχουμε δυσάρεστα νέα για δολοφονίες στο Μεξικό ακτιβιστών ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κύριου Γιώκολα από τη Φιλανδία και Μπέτη Καρίνο Τροίγιο, που σκοτώθηκαν και οι δύο κατά μία αποστολή για τα ανθρώπινα δικαιώματα εκεί. Εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, λοιπόν, θέλω να στείλω συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Είναι σαφές ότι εξακολουθούμε να έχουμε τέτοια θύματα ανά τον κόσμο. Επίσης, πήγα την προηγούμενη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον, όπου εγκαινιάσαμε το γραφείο μας σύνδεσης με το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών. Είχα και συζητήσεις για τις οικονομικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Ηνωμένε Πολιτείες Μιλήσαμε για στρατηγική φύσεως εταιρική σχέση. Και οι συζητήσεις που έγιναν μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας στο Κοινοβούλιο εγκρίνουν τέτοιες σχέσεις με τις Ηνωμένε Πολιτείες επί ίσης ώρες. Τρίτον, 9 Μαΐου θα έχουμε την 60 επέτειο από τη δήλωση Σούμαν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει Open Days Day, δηλαδή μια ημέρα όπου θα μπορεί ο κόσμος να επισκεφθεί το κτίριό μας στο Στρασβούργο. Και στο Λουξεμβούργο, στις Βρυξέλλες το Σάββατο. Ο, η αντιπρόεδρος, ο αντι, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και υπουργοί από την Γερμανία και την Αυστρία θα πάνε στο Λουξεμβούργο. Επόμενο θέμα στην για διάταξη είναι κοινή συζήτηση. με έκθεση του κυρίου Μέντες Δεβίγο που αναφέρεται στην ε, σύγκληση συνέλευσης για την αθεώρηση των συνθήκων και μεταβατικά μέτρα που αφορούν τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ξεκινήσω με τον Ρίλκε, τον ποιητή. Ήταν ο αγαπημένος ποιητής του Δημήτρη Τσάτσου ο οποίος χάθηκε πριν από λίγες μέρες. Εδώ, σε αυτό το χώρο, ο Δημήτρης Τσάτσος και εγώ, στον ίδιο χώρο, παρουσιάσαμε την πρότασή μας για τη συνθήκη του Άμστερνταμ. Και εκεί, για τη σεθήκη του Άμστερνταμ δηλαδή, προτείναμε, εκείνος και εγώ, ό,τι αναθεώρηση γίνει για τις συνθήκες στη συνέχεια να προετοιμαστεί από πριν μέσω της σύγκλησης μιας συνέλευσης. Αυτό είχαμε προτείνει, την κοινοτική μέθοδο, με συνέλευση, που χρησιμοποίησαμε και για να ετοιμάσουμε και την Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και τη Συνταγματική Συνθήκη. Θυμάμαι τον Δημήτρη Τσάτσο, όταν είχαμε προχωρήσει με την ε, διαδικασία αυτή και τον θυμάμαι και τώρα που μιλάμε για την πρώτη αναθεώρηση. Είναι μια πρώτη αναθεώρηση λοιπόν της συνθήκης τη Λισαβόνα αυτή που έχουμε μπροστά μα σήμερα που μιλάει για την τροποποίηση του πρωτοκόλου που όμως συνοδεύεται από μια ανομαλία κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή έγιναν τον Ιούνιο που μας πέρασε οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν δεν είχε ακόμα αρχίσει να ισχύει η συνθήκη της Λισαβόνας. Στις εκλογές λοιπόν εκείνες χρησιμοποίησαμε το καθεστώς που προβλέπει η συνθήκη της νίκαιας, η οποία συνθήκη της νίκαιας δεν μιλάει για 751 ευρωβουλευτές όπως λέει η συνθήκη της Λισαβόνας. Έτσι λοιπόν η εντολή των ευρωβουλευτών ισχύει 5 χρόνια σύμφωνα με την συνθήκη αυτή. Πράγμα που σημαίνει ότι τους 751 δεν μπορούμε να τους έχουμε γιατί υπάρχουν τρεις ευρωβουλευτές από χώρα που χάνει τρεις ευρωβουλευτές που τους έχει εκλέξει και δεν μπορούμε να τους διώξουμε κατά τη διάρκεια της θητείας. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να τροποποιήσουμε το πρωτόκολλο 36 ώστε οι συμφωνίες της Λισαβόνας να αρχίσουν να ισχύουν. Έτσι, κατά τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας, 2009-2014 δηλαδή, που θα αρχίσει να ισχύει η τροποποίηση του πρωτοκόλλου 36, εκτάκτος θα έχουμε 744 ευρωβουλευτές. Σας έστειλε επιστολή, Πρόεδρε, με την οποία σας ζήτησα ότι βάσει το άρθρο 48 της αθήκης να αποφανθεί το Κοινοβούλιο μας επί δύο θεμάτων. Πρώτον, χρειάζεται συνέλευση για να ετοιμάσουμε την τροποποίηση του πρωτόκολλου 36. Δεύτερο ερώτημα. Οι κυβερνήσει, οι ηγέτε κατών και κυβερνήσεων μπορούν να συγκαλέσουν διακυβερνητική διάσκεψη για να τροποποιηθεί το πρωτόκολλο 36. Βέβαια είναι αλληλένδετε οι δύο αυτέ ερωτήσει, παρόλο που τι χειρίζομαι σε δύο διαφορετικέ εκθέσει. Θα ξεκινήσω από το πρώτο, τη σύγκληση τη διακυβερνητική ε, διάσκεψη. Πρόκειται για την εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας βάσει πολιτικής συμφωνίας. Πρόκειται για μια μεταβατική λύση που εκτάκτο χρησιμοποιούμε και η οποία θα λάβει χώρα για τη θητεία αυτή. Η διακυβερνητική αυτή διάσκεψη τι θα κάνει ουσιαστικά θα εφαρμόσει κάτι το οποίο έχουμε ήδη συμφωνήσει για τους 18 αυτούς ευρωβουλευτές, δηλαδή από 12 διαφορετικές χώρες που θα προσθεθούν εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται συζήτηση, Πρόεδρε. Νομίζω ότι η διακυβερνητική διάσκεψη μπορεί να συγκληθεί πάρα πολύ γρήγορα και να λήξει μέσα σε ένα πρωινό γιατί η πολιτική απόφαση έχει ήδη ληφθεί. Γι' αυτό λοιπόν κύριε Πρόεδρε, μα έξι λεπτά μου είπατε ότι έχω, τέσσερα συν δύο. Α, μετά τη συζήτηση. Καλώς. Τότε το μόνο που θα πω είναι ναι στη διακυβερνητική διάσκεψη και Κατά τα άλλα, δεν πιστεύω ότι χρειάζεται να συγκληθεί συνέλευση για ένα θέμα το οποίο έχει εκ των προτέρων λυθεί. Ε, συγγνώμη που έκανα λάθο. Νόμιζα ότι είχα 6 λεπτά και 6 λεπτά ποτέ δεν είχα στη διάθεσή μου εδώ. Οπότε ενθουσιάστηκα. Εν πάση περιπτώσει, ωραία, νομίζω ότι είναι σαφή η θέση μου. Ω εισηγητή, λέω ότι πρέπει να είμαστε υπέρ τη ε, διακυβερνητική ε, διάσκεψη και κατά τη σύγκληση νέα συνέλευση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ συνάδελφε για την έκθεσή σας και για την εισήγησή σας. Θα ήθελα να πω ότι πρόκειται για έξι λεπτά όλα μαζί και περιμέναμε να μιλήσετε δύο λεπτά στο τέλος της συζήτησης. Το είχαμε χωρίσει δηλαδή σε τέσσερα λεπτά στην εισήγηση και δύο στο τέλος ως συμπέρασμα. Δηλαδή ενάμιση σας έμεινε για το τέλος. Λυπάμαι. Αλλά εντάξει, αν έτσι και αλλιώ δύο λεπτά. Συμφωνώ να ζητήσω τώρα εξ στο του Συμβουλίου τον Υπουργό Διέγκο Λόπες Γκαρίντο να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκδηλώσω την ικανοποίησή μου το γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δια του αγαπημένου φίλου και συναδέλφου Ίνιγκο Μέντες Δεβίγο συμπίπτει με την άποψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υπό την εξή έννοια. Η αναθεώρηση του πρωτοκόλου 36, όπως προτείνεται, είναι εκ των ουκ άνευ. Εκ των ουκ άνευ, μιλώ για τη συνθήκη της Λισαβόνας, για να μπορέσουν στο Κοινοβούλιο να έρθουν πριν τις επόμενες ευρωεκλογές ο ρυθμός εκείνος των βουλευτών που ε, κανονικά θα έπρεπε να είναι ήδη παρόντες εάν ε, ίσχυε ε, πριν τις ευρωεκλογές η συνθήκη της Λισαβόνας. Και επειδή είναι λοιπόν μικρή αυτή η αναθεώρηση, δεν χρειάζεται να συγκληθεί συντακτική συνέλευση. Το παράδοξο εδώ ποιο είναι. Ο κύριος Μέντες Δεβίγο και εγώ ήμασταν μέλη της συνέλευσης τότε που συνέταξε σύνταγμα για την Ευρώπη. Και τώρα ε, θα πρέπει να αποφύγουμε αυτή την εξέλιξη γιατί είναι πάρα πολύ μικρή η τροποποίηση αυτή. Και ουσιαστικά είναι μάλλον τυπικό ε, θέμα, διεκπαιρεωτικό ε, στη συνθήκη της Λισαβόνα. Και χαίρομαι που με τον τρόπο αυτό, αν εγκρίνει το Κοινοβούλιο την πρόταση που κάνει ο εισηγητής, κ. Μέντες Δεβίγο, θα μπορέσουν να έρθουν το συντομότερο μετά τη διακυβερνητική διάσκεψη ή ε, νέοι βουλευτές. Και βεβαίως αφού κυρωθούν αναλόγως και στα 27 κοινοβούλια αυτές οι αποφάσεις. Να μπορέσουν να ενταχθούν ε, άλλοι 18 βουλευτές, άνδρες και γυναίκα, ε, από 12 χώρες. Να σας πω ποιες χώρες. Ηνωμένο Βασίλειο, Σλοβενία, Πολωνία, κάτω χώρες. Μάλτα, Λετωνία, Ιταλία, Βουλγαρία, Σουηδία ε, Γαλλία, Αυστρία και Ισπανία. Οπότε οι ε, πολίτες αυτών των χωρών θα ε, είναι σε θέση να έχουν ακόμα καλύτερη εκπροσώπηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ ικανοποιητική η εξέλιξη αυτή η έκθεση με στη Βίγο. Εγκρίθηκε στη Συνταγματική Επιτροπή του Κοινοβουλίου και ελπίζω να εγκριθεί και στην Ολομέλεια με ευρεία πλειοψηφία και το συντομότερο να μπορέσουμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υποδεχθούμε τους 18 νέους βουλευτές που πραγματικά ε, λείπουν από το Κοινοβούλιο αν θέλει να είναι σύμφωνο με τις συνθήκες της Αβώνας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Um, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Διέγκο Λόπες Γαρίδο, εξ του Συμβουλίου, για τη δήλωσή σας ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Μάρος Σεφτσοβιτς, εξ ονόματος της Κομισιόν. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μέντες Δεβίγκο για την εξαιρετική του έκθεση και είμαι ευτυχή που μπορώ να ενημερώσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί η Κομισιόν, για το ότι η Κομισιόν ενέκρινε μια θετική γνωμοδότηση για την έναρξη μιας διακυβερνητικής διάσκεψης μετά από την πρόταση των Ευρωβουλευτών. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε ε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε γνωμοδότηση από την Κομισιόν σε σχέση με αυτό και επειδή πρόκειται για μία μόνιμη πολιτική συμφωνία, το να μπουν δηλαδή σε, να, αναλάβουν καθήκοντα 18 ε, ευρωβουλευτέ όσο γίνεται πιο σύντομα, η Κομισιόν ενέργησε όσο γινόταν πιο γρήγορα. Υπό το φω αυτή τη πρόταση, τονίζουμε πω η διακυβερνητική θα πρέπει να περιοριστεί και να ασχοληθεί με το θέμα των επιπλέον ευρωβουλευτών. Και με χαρά είδα ότι η έκθεση του κ. Μέντες Δεβίγο υποστηρίχθηκε από, από μεγάλη πλειοψηφία στην Επιτροπή ΑΦΚΟ και ελπίζουμε ότι το ίδιο θα συμβεί και αύριο στην ε, ψηφοφορία Τη Ολομέλειας. Ε, να εκφράσω επίσης την ευχή της Κομισιόν ότι η περιορισμένη αλλαγή της συνθήκης που θα συζητηθεί από τη διακυβερνητική θα, είναι σύντομα, θα συζητηθεί σύντομα, θα επικυρωθεί σύντομα και έτσι οι επιπλέον 18 ευρωβουλευτές να αναλάβουν τα καθήκοντά τους όσο γίνεται πιο γρήγορα. Σας ευχαριστώ. για την παρουσίαση τη θέσης της Κομισιόν. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι εδώ μιλάμε για δύο εκθέσεις του συναδέλφου Μέντες Δεβίγκο πρώτα, δηλαδή αναθεώρηση της, των συνθηκών μέτρα σχετικά με την σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η δεύτερη αφορά τη σύγκληση συνέλευση για την αναθεώρηση των συνθηκών για τα μεταβατικά μέτρα που αφορούν τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ήθελα αυτό να το θυμίσω, ότι δηλαδή πρόκειται για κοινή συζήτηση δύο εκθέσεων. Και όπως είπε ο συνάδελφος Νίγκο, Αυτή ήταν και η ερώτηση την οποία απευθύναμε στην Κομισιόν. Τώρα, εξ ονόματος του ΕΛΚ, ο Κάρλο Κασίνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ σύντομα γιατί η Κομισιόν της οποίας ηγούμε έχει φτάσει σε μια ευρεία συνένεση που συμφωνεί με τα όσα ήδη είπατε και άρα δεν χρειάζεται να βαρύνουμε υπερβολικά τη συζήτηση. Το πρόβλημα που υπήρχε και επί το οποίο συζητήσαμε στην Κομισιόν αφορούσε κυρίως το εξή. Ότι δηλαδή τόσο η εκλογική πράξη του 76 όσο και η συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπουν ότι, προβλέπουν ότι άμεσα από τους λαούς εκλέγονται οι ευρωβουλευτές άμεσα από τους λαούς των διαφόρων κρατών. Και εδώ είναι ένα πρόβλημα γιατί τα, τα εκλογικά συστήματα με, οποία, με βάση τα οποία εξελέγησαν οι ευρωβουλευτές αυτές τι θητείε δεν επιτρέπουν να μπουν στο κοινοβούλιο υποψήφοι που είχαν επιτυχία, όχι και απόλυτη, αλλά τέτοια επιτυχία που να μπορούν να μπουν στο Ευρωκοινοβούλιο. Α, κάποια ηλεκτρονικά συστήματα το επιτρέπουν και άλλα όχι. Άρα λοιπόν θα πρέπει να, να τρέξουμε, αν δεν θέλουμε να καθυστερήσουμε πάρα πολύ την ε, ε, ολοκλήρωση του Κοινοβουλίου σε συστήματα διορισμού ε, που είναι έκτακτα και μεταβατικά όπως προβλέπει το Συμβούλιο. Μετά από μακρές συζητήσεις στην Κομισιόν θεωρήσαμε πως αυτή ήταν η σωστή ε, θέση και συμφωνούμε λοιπόν με τα όσα είπατε. Θα πρέπει να σας πω προσωπικά ότι έχω υποβάλει μια τροπολογία που προέβλεπε τον διορισμό παρατηρητών για τη μεταβατική περίοδο πριν από την εκλογή των νέων μελών του Κοινοβουλίου. Αυτή η τροπολογία είναι ακόμα υποσυζήτηση, αλλά θα πρέπει ίσως να την καταψηφίσουμε ακόμα και είναι δική μου τροπολογία, γιατί η συμβαστική τροπολογία προβλέπει μία ε, γρήγορη, άμεση ολοκλήρωση του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Για σοσιαλιστές ε, δημοκράτες. Ο Ραμόν Χάουρεγγι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας πω ότι δεν είναι ίσονο σημασία η απόφαση αυτή που θα λάβουμε σήμερα. Καταρχάς, αναθεωρούμε τη συνθήκη. Για πρώτη φορά τη συνθήκη που πρόσφατα τέθηκε σε ισχύ. Την αναθεωρούμε. Και αυτό δεν είναι κάτι το ευκαταφρόνητρο. Και το δεύτερο που κάνουμε είναι ότι υλοποιούμε τη δυνατότητα αυτή 18 βουλευτέ, που θα είχαν το δικαίωμα να είναι βουλευτέ, ακριβώς αν είχε εγκριθεί πριν τι εκλογέ η συνθήκη και 12 χώρες που έχουν το δικαίωμα να έχουν ε, νέα εκπροσώπηση στο Κοινοβούλιο, γιατί έχει συμφωνήσει το Σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν περισσότερους βουλευτές από όσους ε, διαθέτουν σήμερα για να μπορούν να ασκήσουν αυτό το δικαίωμα. Περί αυτού πρόκειται μόνο, αλλά ε, και αυτό είναι σημαντικό ζήτημα. Ωστόσο, για την αναθεώρηση της συνθήκης. Η συνθήκη ίδια ζητάει ε, να συγκληθεί η συντακτική συνέλευση. Και το Συμβούλιο μας λέει, μα τώρα χρειάζεται συνέλευση για αυτό το πράγμα, για να κυρωθεί μια συμφωνία όλων των χωρών της Ένωσης. Και αυτό που απαντάει το Κοινοβούλιο είναι ότι ε, ναι, δεν χρειάζεται να συγκληθεί σε αυτή την περίπτωση συντακτική συνέλευση και αναθέτει λοιπόν την εντολή στο Συμβούλιο να συγκαλέσει πλέον όχι συνέλευση αλλά διακυβερνητική διάσκεψη για να ε, ξαναρχίσει η διαδικασία αυτή και 27 χώρες να κυρώσουν την αλλαγή και να έρθουν οι 18 βουλευτές που λείπουν και οι 12 χώρες να έχουν την πλήρη τους εκπροσώπηση σύμφωνα με τη συνθήκη. Περί αυτού πρόκειται. αναγνωρίζω ότι είχαμε κάποια δυσκολία ε, όταν χρειάστηκε να εξακριβώσουμε αν ε, θα έπρεπε να εκλεγούν με ευρωεκλογέ οι 18 αυτοί με άλλο τρόπο. Γιατί ανέκυψε αυτό το πρόβλημα. Και θα πρέπει να το δούμε ε, κατάματα. Λύθηκε όμως με τρόπο ικανοποιητικό και Θέλω να ευχαριστήσω όχι μόνο τον εισηγητή της έκθεσης αυτή, τον Μέντας Δεφίγο, αλλά και τον κύριο Νταφ, γιατί καταφέραμε οι τρεις πολιτικές ομάδες μια συμφωνία που κατά την άποψή μου είναι πολύ σημαντική. Τι λέγουμε λοιπόν, ότι ναι, να αναθεωρηθεί αυτή η συνθήκη χωρίς ε, συνέλευση και ταυτόχρονα το Κοινοβούλιο θυμίζει στα εθνικά κοινοβούλια ότι θα πρέπει να αποστείλουν εκλεγμένους, άμεσα εκλεγμένους βουλευτές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και εμείς θα αναθεωρήσουμε στο Κοινοβούλιο μας το ε, ε, ευρωπαϊκό εκλογικό σύστημα έτσι ώστε ε, στην Ευρώπη να έχουμε ένα σύστημα ενιαίο υπερεθνικό για να εκλέγουμε ευρωβουλευτές. Αυτά τα δύο λέμε επίσης και έτσι έχουμε μια ισορροπία πλέον και χαίρομαι πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Άντρου Ντάφ από τους Φιλελεύθερους Δημοκράτες. Ε, αν η συνθήκη είχε αρχίσει να ισχύει νωρίτερα, μια τέτοια πρόταση ε, είχε γίνει, δεν θα τη δεχόμασταν. Το Κοινοβούλιο δεν θα μπορούσε να δεχτεί το γεγονός ότι η Γαλλία θα προσπαθούσε να διορίσει βουλευτές από την Εθνοβουλή στο Ευρωκοινοβούλιο. Και αν τον συμφωνήσαμε μετά από την έναξη ισχύω της ε, συνθήκης, θα είχαμε παραβιάσει τη συνθήκη. Γιατί η πρόταση αυτή δεν σέβεται την αρχή της μειούμενης αναλογικότητας. Δεχόμαστε λοιπόν μια μεταβατική λύση. Η αντιπαράθεση αυτή εκτέθεσε τα προβλήματα που αφορούν τη σύνθεση του Κοινοβουλίου και την εκλογική διαδικασία και με χαρά Διαπιστώνω πως όλες οι ομάδες συμφωνούν πως χρειάζεται ουσιαστική μεταρρύθμιση της εκλογικής διαδικασίας. Το Κοινοβούλιο σύντομα θα υποβάλει προτάσεις που θα απαιτήσουν την σύγκληση μιας διακυβερνητικής διάσκεψης που θα προετοιμαστεί από μια συνέλευση που θα συμπεριλαμβάνει τα εθνικά κοινοβούλια. Με συμμετοχή δηλαδή των εθνικών πολιτικών κομμάτων ώστε να προετοιμαστούμε εγκαίρως για το 2014. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων για τους συναδέλφους στους συναδέλφους για τις ε, επικοδομητικές διαπραγματεύσεις. όσον αφορά την αναθεώρηση της εκλογικής διαδικασίας του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα εξ το των Πρασίνων, ο συνάδελφος Χέφνερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ευρία είναι η συνένεση του θέματος αυτού στο Κοινοβούλιο. Χαιρόμαστε που θα αυξηθεί και ο αριθμό των μελών του Κοινοβουλίου και θα υποδεχθούμε 18 νέα μέλη. Και τώρα θέλουμε να δημιουργήσουμε τι προποθέσει να έρθουν εδώ οι άνθρωποι αυτοί και να μπορούν να συνεργάζονται μαζί μα. Υπάρχει όμω μια μικρή διαφορά που ε, στην ουσία είναι πολύ μεγάλη. Γιατί έχει να κάνει ε, με τη βάση της εργασίας μας αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την αρχή της δημοκρατίας και τη λειτουργία του κοινοβουλίου του ίδιου. Και ποιο είναι αυτό. Ποιος αποφασίσει ποια θα είναι αυτά τα νέα μέλη. Και αυτό είναι ένα θέμα κεντρικό. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, λέει η συνθήκη, εκλέγονται για μία πενταετία σε μία άμεση καθολική και μυστική ψηφοφορία από τους πολίτες. Σε 11 από τα 12 κράτη έγινε αυτό και μια χώρα λέγει ότι αν δεν γίνονται αυτά τα πράγματα να στείλουμε βουλευτές άλλους που έχουμε άλλους βουλευτές αλλά είναι εκλεγμένοι για τελείως διαφορετική δουλειά από τους ε, πολίτες. Αυτό ε, ε, παραβιάζει την αρχή της δημοκρατίας ε, και θα μπορούσαμε, αν ήταν απλώς τεχνικό το ζήτημα, να μην κάνουμε καθόλου συνέλευση. Αλλά πρέπει να τηρηθεί η συνθήκη. Εδώ κινδυνεύει η συνθήκη να παραβιαστεί. και αυτό εμείς επιμένουμε να γίνει συνέλευση, που είναι καταπληκτική μέθοδος ακριβώς σε τέτοια θέματα, να επιτυγχάνει κανείς συνένεση στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. E, Ευχαριστούμε. Εκ μέρους των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών, ο κύριος Φόξ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι για την έκθεση αυτή και για την ανάγκη που εκφράζει για μια συνέλευση η οποία θα ξόδευε δίκως τα χρήματα του φορολογούμενου. Δεν χρειάζεται. δεν χρειάζεται να συζητηθεί τίποτα παραπάνω για ολοκλήρωση. Τουλάχιστον έτσι πιστεύουν όσοι βρίσκονται στη δικιά μου εκλογική περιφέρεια. Κάθε άλλο. Ναι, μεν, χαίρομαι για τα μέτρα που θα επιτρέψουν σε 18 νέου ευρωβουλευτέ να έρθουν εδώ, αλλά από την άλλη μεριά δεν νομίζω ότι πρέπει να έχουν το καθεστώ του παρατηρητή μέχρι να αρχίσουν να ισχύουν τα μεταβατικά μέτρα. Γιατί τότε θα έπρεπε να ζητούν αποζημιώσει και μισθού χωρίς να είναι σε θέση να ψηφίζουν, χωρίς να έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν. Γι' αυτό λοιπόν και πιστεύω ότι όλη η συζήτηση είναι λάθος. Γιατί ενώ προσπαθούμε να κάνουμε περικοπές στις δημόσιες ε, δαπάνες και το ζητάμε αυτό από όλε τις χώρες, ε, πρώτα απ' όλα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να δώσει το παράδειγμα για το πώς ξοδεύει τα χρήματα του φορολογουμένου. Θα καταψηφίσουμε λοιπόν την έκθεση αυτή, γιατί δεν δίνει σημασία σε αυτήν την τόσο βασική για μένα αρχή. Ευχαριστούμε, συνάδελφε τώρα εκ μέρους της Ευρωπαϊκής ε, Ενωτικής Αριστεράς, ο κύριος Ζόντεγκάρτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, είμαι σίγουρος ότι δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε παρά που διαφωνούμε για πολλά θέματα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εδώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι υπάρχουν κάποιες ανησυχίες. Πρώτα απ' όλα, πώς χαίρει νομιμότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με αυτή τη διαδικασία, αν δεν ε, εκλέγονται με καθολική ψηφοφορία οι νέοι αυτοί βουλευτές. Υπάρχει μια πρόταση που προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση, που σημαίνει ότι τα επόμενα τέσσερα χρόνια θα υιοθετούμε μέτρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και που θα τα έχουν υιοθετήσει άνθρωποι οι οποίοι δεν θα έχουν εκλεγεί με καθολική ψηφοφορία. Αυτός είναι ο λάθος τρόπος. Είναι μια ατυχής εξέλιξη αυτή. Και γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξει η συνθήκη, αλλά και στην πράξη. Όταν η Ρουμανία και η Βουλγαρία εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2007, για δυόμιση χρόνια δεν μπορούσαν να έρθουν εδώ ευρωβουλευτέ χωρί εκλογέ. Κάνανε εκλογέ και μετά στείλανε εδώ ευρωβουλευτέ. Αυτό πρέπει να γίνει και τώρα. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ο κύριο Μάσερσμιτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπάρχει κάτι περίεργο εδώ για αυτή την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Για χρόνια έχουμε ακούσει ότι η συνθήκη της Λισαβόνας αποτελεί το μέσο με το οποίο έχουμε δημοκρατία και διαφάνεια που είναι υπέρ των πολιτών και τώρα στην πρώτη του θητεία μετά τη Λισαβόνα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι σαν να λέει όχι στην καθολική ψηφοφορία, όχι σε αυτά τα οποία συζητήσαμε τα τελευταία χρόνια για το γιατί θέλαμε τη συνθήκη της Λισαβόνας. Κάτι παράδοξο συμβαίνει εδώ, δεν νομίζετε. Εμείς πρέπει να πάρουμε στα σοβαρά τις υποσχέσεις που κάναμε στους πολίτες. Για το ότι δηλαδή με καθολική ψηφοφορία εκλέγοντος ή έρχονται εδώ. Και όχι άνθρωποι που εκπροσωπούν κυβερνήσεις, αλλά άνθρωποι που εκπροσωπούν τους πολίτες που τους ψηφίζουν. Αυτοί πρέπει να εδρεύουν εδώ. Πράγμα το οποίο δεν θα ισχύει εφόσον εγκριθούν οι δύο αυτές εκθέσεις. Το όλο επιχείρημα που στήριξε τη συνθήκη της Λισαβόνας είναι κάτι το οποίο πετάμε στα σκουπίδια με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορώ και ούτε και ο τόσο πρόεδρος ομάδας θα μπορούσε να εγκρίνει κάτι τέτοιο. Ευχαριστούμε. Και τώρα, εκ μέρους των μη εγγεγραμμένων, ο κύριος Γκόλνης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα πάω κατευθείαν στο θέμα μας. Το άρθρο 2 της έκθεσης του αδέλφου Μέντες Δεβίγο σωστά τονίζει το γεγονός ότι μία από τις προτάσεις του Συμβουλίου άμεσα αντιτίθεται με ε, το πνεύμα της πράξης του 1976 και είναι ο διορισμός από τα Εθνικά Κοινοβούλια ε, Ευρωβουλευτών. Σύμφωνα με την πράξη του 1976 θα πρέπει να έχουν εκλεγεί με άμεση καθολική ψηφοφορία. Όσο και αν αγαπώ τον εισηγητή, λυπάμαι που δεν λαμβάνει περισσότερο και πιο αυστηρά και ξεκάθαρα στο άρθρο 5 αυτή την αρχή. Εάν τα κράτη δεν θέλουν να κάνουν ε, συμπληρωματικές εκλογές, αρκεί να ληφθούν υπόψη ε, τα αποτελέσματα των εκλογών του 2009 και να εξισωθούν ε, στη συνέχεια ε, με τους νέους βουλευτές, να γίνει ένας συμψηφισμός ε, και να οριστούν οι νέοι βουλευτές σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών. Οτιδήποτε διαφορετικό θα ήταν κατά της δημοκρατίας. Ιδιαίτερα στη χώρα μου, όπου η Εθνοσυνέλευση δεν εκλέγεται με τρόπο αναλογικό και θα ήταν κυβερνητικός διορισμός αυτό που αντιτίθεται στο πνεύμα των συνθήκων. Μάριο Μάουρο, Μάριο Μάουρο, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, παραμένει μυστήριο το γεγονός ότι το Συμβούλιο θα μπορούσε να πάρει τόσο ελαφρά ένα τέτοιο ε, θέμα. Εύχομαι ότι αυτή η δυσάρεστη <clears throat> κατάσταση δεν θα αφήσει άσχημα ίχνη ώστε να μην διατρέξει κίνδυνο η αξιοπιστία των θεσμών μας ε, να σας δώσω το συγκεκριμένο παράδειγμα. Η Ιταλία καλείται να εκλέξει έναν βουλευτή σε μια δεχόμενη επιπλέον ε, εκλογική διαδικασία. Όμως ε, είναι δυνατόν να περάσουμε σε εκλογές όπου θα έχουμε μια πιθανότατη προσέλευση όχι πάνω από το 5% των εκλογέων ή μήπως θα έπρεπε να δούμε τις τα τελευταία αποτελέσματα του 2009 για να εγκρίνουμε έναν βουλευτή που έχει εκλεγεί με καθολική ψηφοφορία, καθολικές εκλογές. Σε πάση περιπτώσει δεν μπορεί η Ευρώπη να επιτρέψει τον εαυτό της ε, θεσμικά σφάλματα οι 18 ευρωβουλευτές θα πρέπει ταυτόχρονα να φτάσουν στο Ευρωκοινοβούλιο ώστε να μην ε, ε, διαταραχτεί η λεπτή ισορροπία που υπάρχει ανάμεσα στις διάφορες ε, ομάδες. Πιστεύω ότι είναι αδιανέοητο να μην εκλεγούν οι ευρωβουλευτές αυτοί για το υπόλοιπο της θητείας μέχρι το 2014. Άρα λοιπόν θα πρέπει επιγόντως να εγκριθεί η σύσταση και η σχετική έκθεση ώστε να δοθεί το πράσινο φως στο πρωτόκολλο 36 τη ε, συνθήκης της Λισαβόνας χωρίς να περάσουμε από το εργαλείο της συνέλευσης αλλά προχωρώντας άμεσα όπως προτείνει ο συγχυγητής στη σύγκληση μιας διακυβερνητικής διάσκεψης. Θα πρέπει δηλαδή να ακολουθήσουμε το πιο σύντομο δρόμο γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν και πολλά να πούμε. Δηλαδή θα πρέπει κανονικά να γυρίσουμε σελίδα και να ξαναρχίσουμε με έναν επικοδομητικό ε, τρόπο από, ξεκινώντας από ένα γεγονός πολύ αρνητικό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Γκρό για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή Μέντες Δεβίγο για τη συνέλευση. Πραγματικά ε, δεν έχει νόημα ε, για μια λεπτομέρεια να συγκληθεί ολόκληρη συνέλευση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το 1979 εκλέγεται άμεσα καθολικά και μυστικά και στο μέλλον θα το τηρήσουμε αυτό. Και καλά θα κάναμε και εμείς και το Συμβούλιο να λύσουμε αυτό το θέμα το συντομότερο σε διακυβερνητική διάσκεψη. Διότι 18 συνάδελφοι, άνδρες και γυναίκες, κυρίως οι 16 από τους 18, ε, ε, είναι λίγο μετέωροι και αυτό είναι μια κατάσταση αρκετά αφόρητη. Και το βαλάκι είναι και πάλι στο γήπεδο του Συμβούλιου. Παρακαλώ λοιπόν το Συμβούλιο να το λύσει αυτό και να μην υποκύψει στον πειρασμό σε ένα κράτος μέλος να αφήσει να είναι τα πράγματα θολά και συγκεχημένα. Έχασαν την ευκαιρία που φταίει και αυτή η χώρα που δεν ετέθηκε σε ισχύ νωρίτερα η συνθήκη τη Λισαβόνα. Σε πάση περιπτώσει, είναι καλή η έκθεση Μέντε στη Βίγο ω αφετηρία, αλλά καλά θα κάνει το Συμβούλιο, επαναλαμβάνω, να μην υποκύψει σε αυτό το πειρασμό, να δεχτεί αυτό που λέει μια χώρα, ότι να έρθουν βουλευτέ ενό Εθνικού Κοινοβουλίου ως απεσπασμένη. Γιατί θα είναι και προηγούμενο αυτό. Και εγώ δεν είμαι πρόθυμος να χωρίσω τέτοια προηγούμενα. Υποστηρίζω πλήρως τον εισηγητή με αυτό τον περιορισμό. Όχι εθνικοί βουλευτές. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Μπελιέ για ένα λεπτό. Σα ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Γαλλία είναι το μόνο κράτο μέλο που δεν προέβλεψε την έναρξη ισχύω τη συνθήκη τη Λισαβόνα και αρνείται να στηριχτεί στα αποτελέσματα των ευρωεκλογών του Ιουνίου 2009. Ε, Δεχόμενη την τρίτη εξαίρεση για τη Γαλλία, μας ζητάτε να παραβιάσουμε ένα βασικό στοιχείο του πρωτογενού δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την άμεση δηλαδή εκλογή των Ευρωβουλευτών, από την οποία αντλούμε την νομιμότητά μας εδώ και 31 χρόνια. Θα υποκληθούμε στη βούληση του Συμβουλίου με υπό την πίεση ενός κράτους που εκφράζει μια κάποια περιφρόνηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αρνηθούμε να ε, αλωτριώσουμε την ευρωπαϊκή μας ταυτότητα και την ε, ευρωπαϊκή δημοκρατία. Οι ευρωπαίοι πολίτες είναι που εκλέγουν τους βουλευτές και όχι τα κράτη-μέλη. Δεν θα πρέπει λοιπόν να δεχτούμε παρά μόνο μια συνέλευση που θα προετοιμάσει μια διακυβερνητική και όχι μια απλή διακυβερνητική διάσκεψη. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Κόλμαν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η καθυστέρηση της επικύρωσης ε, του η συνθήκης της Λισαβόνας έμενε ότι 756 βουλευτές αντί για 751 ήταν αυτοί που ορίστηκαν. Αυτό κατέληξε στο να κατανεμηθούν 18 έδρες σε 12 κράτη-μέλη και με την Γερμανία να χάνει τρεις έδρες. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει μια περαιτέρω επιπλοκή είναι ότι η συνθήκη ορίζει το σύνολο των, ε, του αριθμού δεν πρέπει να, των ευρωβουλευτών πρέπει να ξεπερνά του 751. Το να συμπεριληφθούν οι 18 χωρί να απολεστούν οι τρει γερμανικέ έδρε θα απαιτήσει την αναθεώρηση του πρωτοκόλλου 36 τη συνθήκη Λισαβόνα. Αυτό θα πρέπει να γίνει μέσω μια συνέλευση που θα καταλήξει σε προτάσει που θα συμφωνήσουν τα κράτη-μέλη για ενσωμάτωση στη συνθήκη μέσω τη τροποποίηση αυτή. Αν δεν γίνει κατέξατα παράνομη οποιαδήποτε ενέργεια στην οποία θα προβεί αυτό το κοινοβούλιο, με τη βάση δηλαδή των 754 έναντι 751 που είναι το νόμιμο. Πρόκειται για σημαντική μεταρρύθμιση και τροποποίηση τη συνθήκη τη Λισαβόνα που απαιτεί ε, επανεπικύρωση από όλα τα κρατημέλη και θα δώσει τη δυνατότητα σε μεμονωμένα, για μεμονωμένα εθνικά ε, ε, δημοψηφίσματα. Παρακαλώ ε, το σώμα να απορρίψει αυτή την πρόταση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τρεζεσκόσκη για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Διαφωνώ με τον προλαλήσαντα. Το κοινοβούλιο μας καλείται να απαντήσει κατά πόσο θα πρέπει να συγκαλέσουμε συνάλευση για να αποφασίσει όχι. Συγγνώμη, την ε, διακυβερνητική διάσκεψη όχι. Και λέμε ότι ναι, πρέπει να έχουμε τη διακυβερνητική διάσκεψη και ότι με τη συνθήκη της Λισαβόνας ενισχύεται η νομιμότητά μας. Δεν θέτει προηγούμενο για το μέλλον, διότι σημαντικά θέματα που έχουν να κάνουν με τροποποίηση της συνθήκη της Λισαβόνας απαιτούν έτσι κι αλλιώς τη σύγκληση συνέλευσης. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Ίνικο και τους συντονιστές που πήραν την απόφαση που πήραν. Δεν ήταν εύκολο. Είχαμε πρόβλημα με τους 18 ε, καινούριου ευρωβουλευτές, επειδή ορισμένες χώρες μέλη δεν προβλέπουν σχετική διαδικασία. Αποφασίσαμε όμως παρόλα αυτό ότι η αντιπροσωπευτικότητα είναι το πιο σημαντικό θέμα και αυτή είναι η αρχή που πρέπει να μας καθοδηγεί στις αποφάσεις μας. Το σώμα λοιπόν πρέπει να έχει ισορροπημένη εκπροσώπηση από τα κράτη-μέλη και γι' αυτό και οδηγηθήκαμε σε μια πραγματιστική, ρεαλιστική λύση και ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να αποφασίσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα για τον τρόπο με τον οποίο θα επιλέξουν τους νέους ευρωβουλευτές και εννοείται ότι όλοι οι νέοι ευρωβουλευτές θα πρέπει συγχρόνως να έρθουν και κατά προτίμηση με απευθείας εκλογές. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Γκυγιόμ. Τώρα για δύο λεπτά. Παρακαλώ κύριε Γκυγιόμ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Το θέμα των νέων ευρωβουλευτών δεν είναι κάτι καινούριο. Θυμόμαστε ότι και ο συνάδελφος Λαμασούρ είχε δουλέψει πάνω σε αυτό στην προηγούμενη θητεία. Μας εκπλήσει λοιπόν η περίπλοκη προετοιμασία που γίνεται από τη Γαλλία, ιδιαίτερα για τους δύο νέους. Μπορεί κανείς να φανταστεί, ότι, να φανταστεί από πριν ότι κάποια στιγμή θα είχαμε την Λισαβόνα, οπότε κάποια στιγμή το νέο αυτό θέμα θα πρέκυπτε για τους δύο καινούριου ευρωβουλευτές δηλαδή. Γιατί δεν το πρόβλεψε η Γαλλία. Με το πρωτόκολλο 36 η Γαλλία μπορεί να ορίσει ε, στην ε, Εθνοσυνέλευση δύο νέους ευρωβουλευτές αλλά έτσι χάνουμε το βασικό κανόνα που λέει ότι οι ευρωβουλευτές εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία. Αυτός είναι ο όρος για την εκλογή και αυτό είναι πράγμα με το οποίο διακυδεύεται η Διεξοπιστία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Από την άλλη βέβαια οι εκλεγμένοι από τις άλλες 11 χώρες που ορίστηκαν με σωστές διαδικασίες δεν πρέπει να εκβιάζουν την κατάσταση, δεν είναι καλό αυτό, θα πρέπει να έρθουν όσο γίνεται πιο γρήγορα εδώ και να αρχίσουν τις εργασίες τους εδώ αντί να καθυστερούν εξαιτία μιας χώρας. Μία διακυβερνητική θα μπορούσε να λύσει το ζήτημα, αλλά εμείς ζητάμε πάνω απ' όλα η Γαλλία να φροντίσει να λύσει το θέμα όπως έκαναν και οι υπόλοιποι. Είναι απαράδεκτη αυτή η κατάσταση και πλήττει πάνω απ' όλα τους Ευρωπαίους πολίτες. Όλα αυτά όμω μα δείχνουν ότι πρέπει να υπάρχει ένα ομοιόμορφο τρόπο επιλογή των νέων ευρωβουλευτών με άμεση και καθολική ψηφοφορία και αυτό ίσως πρέπει να αποφασιστεί με τη σύγκληση μιας ε, συνέλευσης. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Γκουρμάη, η κυρία Γκουρμάη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, συνάδελφοι. Ευχαριστώ για την δουλειά που έχει κάνει και ευχαριστώ και για τους συναδέλφους που συμμετείχαν. Μετά από πολύ σοβαρά προβλήματα επικύρωσης, η συνθήκη της Λισαβόνας είναι επιτέλους ενισχύ. Θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία Χρειάζονται θεσμικέ μεταρρυθμίσει, αλλά θα πρέπει να ασχοληθούμε με τη λήψη αποφάσεων προ όφελο όλων των Ευρωπαίων ε, πολιτών θα πρέπει να έχουμε αποτελεσματική διαδικασία λήψη αποφάσεων. Οι Ευρωπαίοι θέλουν να κάνουμε τη δουλειά μα αποτελεσματικά και με διαφάνεια. Καλή συνεργασία θέλουν επίση ανάμεσα στα διάφορα θεσμικά οργανά και είμαι σίγουρη ότι η προτινόμενη συμβαστική, ο προτινόμενο συμβιβασμό θα είναι μια βιώσιμη λύση. Πιστεύω πω έτσι θα εξυπηρετήσουμε του Ευρωπαίου πολίτες. Και τέλο. προσωπικά να σα πω ότι ορισμένοι ότι θα εμπλουτιστεί το κοινοβούλιο, θα, θα έχει προσθέμενη αξία το όργανο μας όταν θα έρθουν και οι επιπλέον 18 συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ. Δίνω το λόγο στους ομιλητές που ζήτησαν το λόγο για τη διαδικασία Catch the Eye. Ξεκινάμε με τον κύριο Λεγκρίπ. Κυρία Αλεγκρίπ, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου μετά από άλλους ομιλητές να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον συνάδελφο Μέντες Δεβίγκο που επετέλεσε μια αξιοπρόσεκτη εργασία υπό συνθήκες που κάποιες φορές ήταν ιδιαίτερα εμπαθείς. Το, αυτό συμβαίνει στη Συνταγματική Επιτροπή, στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και στο ύψος της έντασης και του ενδιαφέροντος που έχει βέβαια το Ευρωκοινοβούλιο για τα μεγάλα θέματα που τα αφορούν άμεσα, δηλαδή τη σύνθεση του σώματος και τον τρόπο ορισμού των μελών του Ευρωκοινοβουλίου. Για μια ακόμη φορά ο εισηγητής μπόρεσε να συγκεντρώσει απόψεις και συμβολές που κάποιες φορές ήταν διαφορετικές και να συνοψίσει σε ένα κείμενο εξαιρετικά ισορροπημένο όλες αυτές τις θέσεις. Θέλω να τον ευχαριστήσω και πιστεύω ότι τα όσα αναφέρονται σε αυτές τις δύο εκθέσεις για, την, τα μεταβατικά μέτρα ή και για την σύγκληση διακυβερνητικής διαπνέονται από ρεαλισμό, πραγματισμό και αποτελεσματικότητα. Αυτό περιμένουν οι συμπολίτες μας από την Ευρώπη. Για ένα λεπτό η κυρία Κάλεμπαχ. Ευχαριστώ και εγώ πολύ τον εισηγητή και όλους τους και εισηγητές και πιστεύω ότι ως Κοινοβούλιο σήμερα θα πρέπει να στείλουμε ένα σαφέστατο μήνυμα ότι χαιρόμαστε πάρα πολύ που θα υποδεχθούμε νέους Φιλαδέλφους στο Κοινοβούλιο και να μην δείχνει αμέλεια το Συμβούλιο, να τονίσουμε και πάλι αυτή την εντολή, το συντομότερο να δοθεί λύση για να έρθουν εδώ βουλευτές ελεύθερα εκλεγμένοι, 18 παρακαλώ τον αριθμό, και να πιάσουν δουλειά. Διότι ως κοινοβούλιο δεν έχουμε στόχο να εκπροσωπούμε όσο γίνεται καλύτερα τους πολίτες, αλλά να εργαζόμαστε όσο γίνεται αποτελεσματικότερα στις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Και γι' αυτό περιμένουμε του συναδέλφου για να αξιοποιήσουμε και τη γνώση του. Οι άνθρωποι έχουν εκλεγεί με τρόπο σωστό και όπω πρέπει και ω Αυστριακοί Χαίρομαι πάρα πολύ ε, που θα έρθει ο συνάδελφο ο στο συντομότερο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε δεν πρόλαβε να στεγνώσει το μελάνι ε, της ατυχής σας ε, συνθήκης της ε, Έχουμε τη νέα αναθεώρηση και μιλάμε ήδη για βουλευτές φαντάσματα. Γεγονός είναι αυτό. Γι' αυτό πώς συνέβη. Έχουμε διαφορετικά εκλογικά συστήματα που έχουν και προβλήματα δημοκρατίας εν γενή. Και σε περιφερειακό επίπεδο, ας πούμε, ορισμένοι είναι υποψήφοι και δεν έχουν λίστες τότε δεν είναι πολύ δύσκολο να υπάρχουν επιλαχόντες. Αλλά μιλάμε για εκλογή, όχι επιλογή βουλευτών από εθνικά κοινοβούλια. Και επίσης θα πρέπει να δίνουμε συγκεκριμένες προφορίες για τους βουλευτές, για τη δραστηριότητά τους, για τη δράση τους, για τις αποδοχές τους και να μην έχουμε αυτές τις καταστάσεις φαντασματικές γιατί ε, υπονομεύουν την ε, αξιοπιστία μας στα μάτια των πολιτών και την εμπιστοσύνη των πολιτών. Λοιπόν, να δούμε πότε θα έρθουν οι συνάδελφοι, τι καθεστώ θα έχουν, η συνθήκη τη Σαββόνα, ε, πώς θα τεθεί σε ισχύ, τι θα γίνει όταν μπει η Κροατία. Πολλά ανοιχτά ζητήματα. Περιμένουν ε, γρήγορα ε, δήλωση και εξήγηση οι πολίτες από το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Σικέρσκι. Δεν ξέρω αν το προέφερα καλά. Ένα λεπτό. Ε, όλα αυτά θα έπρεπε να έχουν γίνει πριν από ένα χρόνο με την σύγκληση της διακυβερνητικής. Ε, υπάρχει το ειδικό πρωτόκολλο όσον αφορά τις νέες εντολές. Ε, η συνθήκη πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως και σύντομα. θα πρέπει να θυμίσουμε πως είναι στο συμφέρον των κρατών να αυξήσουν την σύνθεση την, για να, και να επικυρώσουν ώστε ε, τα κρατημέλη να μπορέσουν να παρουσιάσουν γρήγορα τους, εκλο, τους ε, ε, εκλεγμένους τους εκπροσώπους. Είναι θέμα αντιπροσωπευτικότητας και δημοκρατίας για την Ένωση. Άρα λοιπόν όλοι οι βουλευτές θα πρέπει να κληθούν στην ίδια στιγμή ώστε να μην υπάρξει κατηγορία για κακή λειτουργία, δυσλειτουργία του θεσμού μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Τσβέρα. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Αξιότιμε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, Συμβούλιο, Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ε, συναδέρφους που λένε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συμπληρωθεί και να ξεκινήσει τις εργασίες του με πλήρη σύνθεση όσο γίνεται πιο γρήγορα. Εφόσον όμως αλλάζουμε τη συνθήκη και δεν έχουμε εφαρμόσει τις αλλαγές σύμφωνα με τη νέα συνθήκη, αυτό δεν έχει γίνει και πρέπει να γίνει. Είναι ο καλύτερος τρόπος προκειμένου να δώσουμε νομική βάση στο έργο μας. Θέλω να συγχαρώ λοιπόν τον εισηγητή, ο οποίος προσπαθεί να βρει τον καλύτερο δρόμο, την καλύτερη νομική λύση. Η σημερινή συζήτηση δείχνει ότι έχει βρει το σωστό τρόπο για να γίνει αυτό. Είμαι κι εγώ ένας από αυτούς που περιμένει τους νέους ευρωβουλευτές, γιατί πιστεύω ότι τους χρειαζόμαστε εδώ. Αυτοί που δεν φρόντισαν να προβλέψουν με τις προηγούμενες εκλογές ότι θα πρέπει να βρουν, να ορίσουν δύο καινούριους ευρωβουλευτές, έχω να τους πω ότι για τους δύο που δεν θα έχουν ε, εκλεγεί, ε, δεν νομίζω ότι αυτό θα πλήξει την νομιμότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο τελευταίος ε, που ζήτησε το λόγο για ένα λεπτό, ο κύριος Κέλλη. Όπως και οι συνάδελφοι, πιστεύω πως ε, αυτοί που εκλέγονται στο Ευρωκοινοβούλιο έχουν ε, το δικαίωμα να πάρουν τις έδρες τους, όπως και οι 736 ευρωβουλευτές που έχουν πάρει τις έδρες τους τελευταίους 12 μήνες. Είναι ένα πολύ, πολύ κέριο ζήτημα που χρειάζεται και μια κέρια λύση, γιατί σε τέσσερα χρόνια θα έχουν όλα καταλαγιάσει και θα λειτουργούν όμαλα. Επίσης είναι λάθος που κατηγορούμε τα κρατη που δεν προέβλεψαν 12 μήνες πριν και δεν ε, ανέλαβαν δράση. Πριν από 12 μήνες υπήρχαν πολύ μεγάλε πιθανότητε να μην επικυρωθεί η συνθήκη τη Λισαβόνα και σίγουρα αυτή ήταν η θέση που πολλοί στη χώρα μου υποστήριζαν. Τώρα όμω που έχει επικυρωθεί είναι σημαντικό οι άνθρωποι που έχουν εκλεγεί να μπορέσουν να πάρουν τι έδρε του και να συμβάλλουν μέχρι τι επόμενε εκλογέ, σε τέσσερα χρόνια όπου όλα θα είναι ομαλά πια και θα έχουν ρονταριστεί. Grazie. Ε, diamo ora ε, E Ευχαριστώ. Και τώρα το Συμβούλιο. Παρακαλώ, κύριος Λόπες Καρίδο. Ευχαριστώ. Θέλω να πω ότι συμφωνώ με εκείνους από εσά που υπογράμμισαν πόσο σημαντικό είναι να λυθεί αυτό το θέμα που βρίσκεται σε κρεμότητα βάσει της ηθίκης της Λισαβόνας. Οι 18 δηλαδή αυτοί οι ευρωβουλευτές, γυναίκες και άντρες, που πρέπει να προσθεθούν. Διότι οι προηγούμενες εκλογές έγιναν, βλέπετε, λίγο πιο πριν από την έγκριση της ηθίκης της Λισαβόνας. Χρειάζεται λοιπόν τροποποίηση του πρωτοκόλου 36. Και συμφωνώ επίσης απόλυτα με εκείνους οι οποίοι εξέφρασαν την άποψη για το ότι αυτό πρέπει να γίνει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Διότι η απουσία των ευρωβουλευτών αυτών, ανδρών και γυναικών, από το σώμα, που εκπροσωπούν πολίτες από 12 ευρωπαϊκές χώρες, είναι κάτι που πρέπει να προχωρήσει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Γι' αυτό λοιπόν και συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Μέντες Δεβίγο, που προτείνει να μην συγκληθεί συντακτική συνέλευση, και να συγκληθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα μια νέα διακυβερνητική, ώστε όσο γίνεται πιο γρήγορα να γίνουν οι τροποποίησεις που χρειάζεται στα κράτη-μέλη και να έχουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα τους νέους 18 ευρωβουλευτές που θα έπρεπε κανονικά να είναι εδώ από την αρχή της τρέχουσας θητείας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και τώρα το λόγο έχει η Κομισιόν. Παρακαλώ κύριε Επίτροπε Σεύκοβιτς. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω πως και αυτή η συζήτηση απέδειξε πως προσπαθούμε να λύσουμε την έκτακτη αυτή κατάσταση και αναζητούμε μια ρεαλιστική και πρακτική λύση και, ε, μεταβατική, για τη μεταβατική αυτή περίοδο και γι' αυτό και καλωσορίζω την ε, πολύ ρεαλιστική προσέγγιση του, κυρία, του κυρίου Μέντες Δεβίγκο και την έκθεση που έχει προετοιμάσει και από την αίσθηση που πήρα από την συζήτηση υποστηρίζεται από το σώμα. Γιατί κοινό ο στόχο μα είναι να έχουμε 18 νέου ευρωβουλευτέ όσο γίνεται πιο σύντομα. Και να επανέλθουμε στην θέση της Κομισιόν και μας, ρωτη... μας ρωτήσατε απευθείας την ερώτηση για το πώς θα πρέπει να διαχειριστούμε αυτή την αλλαγή. Με ποια μέσα. Και η Κομισιόν συμφώνησε ξεκάθαρα με την ε, διακυβερνητική λόγω του φύση και του εύρου της αλλαγής που θα συζητηθεί. Τώρα, θέλουμε να μιλήσουμε για το πώς θα επιλεγούν οι επιπλέον βουλευτέ. Ε, σίγουρα αυτό θα θυγεί στο πλαίσιο τη διακυβερνητική διάσκεψη. Αλλά να προσθέσω επίση ότι όταν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέταζε αυτό το θέμα, ήταν ξεκάθαρο πως το Συμβούλιο προσπαθούσε να βρει μια ισορροπία. Μια ισορροπία ανάμεσα στη φυσική επιθυμία αυτοί οι βουλευτές να επιλεγούν όσο γίνεται πιο κοντά στις ευρωεκλογέ για το Κοινοβούλιο και την ανάγκη για εθνικές ρυθμίσεις. Και γι' αυτό είχαμε αυτές τις τρεις επιλογές, για να καλύψουμε την πραγματικότητα της σημερινής κατάστασης, η οποία φυσικά θα ε, τακτοποιηθεί στις επόμενες εκλογές. Επίσης, να καλωσορίσω τις εσωτερικό, τον εσωτερικό προβληματισμό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο σε σχέση με τις μελλοντικέ αλλαγές για τις ευρωεκλογές να υπογραμμίσω ότι όλα αυτά παραμένουν διαφορετικά ζητήματα από αυτά που συζητάμε σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Για να κλείσουμε τη συζήτηση, το λόγο έχει ο κύριος Μέντες Δεβίγο. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, όταν από διαφορετικές και αποκλίνουσες θέσεις Κόλμαν, Μάουρο ή Γκόλνης καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η εκλογή των Ευρωβουλευτών και τα εκλογικά συστήματα είναι προβληματικά, αυτό σημαίνει, κυρία Πρόεδρε, ότι χρειαζόμαστε ε, μια ενιαία ομοιόμορφη εκλογική διαδικασία. Αυτό είναι από τη συνθήκη της Ρώμης εντολή που έχουμε. Οπότε θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους ε, ε, και τους συνεισηγητές και τον κύριο Χάουρη και ε, Νταφ. Συμφωνήσαμε για τροπολογία αύριο, ελπίζω να υπερψηφιστεί από το Κοινοβούλιο έτσι ώστε το θέμα αυτό, το ζήτημα της νέας εκλογικής διαδικασίας για την εκλογή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λυθεί σύντομα. Και έτσι νομίζω θα διασκεδάσουμε οποιασδήποτε ανησυχίες τέτοιου τύπου. Ο κύριος Σαρκόσκι μίλησε για την ε, απαραίτητη αντιπροσωπευτικότητα του Κοινοβουλίου. Μα αυτό το είπαν και πολλοί ε, προλαλήσαντες. Κατέστη σαφέστατο. Και ε, συμφωνώ, το λέμε και στην έκθεση, στο πρώτο άρθρο, οι 18 να έρθουν όλοι μαζί. Αλλιώς ακριβώς τα χάναμε σε αντιπροσωπευτικότητα. Και για να έρθουν όλοι μαζί, για να γίνει αυτή η πολιτική δικαιοσύνη στη ε, συνθήκη της Λισαβόνας θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Γιατί έκτακτες και μεταβατικές περιστάσεις απαιτούν και μεταβατικές και έκτακτες λύσεις. Εγώ δεν σας κρύβω ότι δεν μ' αρέσει αυτή η δυνατότητα να έρθουν εδώ βουλευτές που να μην έχουν βγει από τις εκλογές του 2009. Το λέω με κάθε σαφήνεια. Και στην παράγραφο 2. Εάν θα πρέπει να επιλέξω μεταξύ αυτού και να μην έρθουν καθόλου οι 18 ή θα βρούμε άλλη λύση ή θα έρθουν οι 18 και θα ε, είμαστε σύμφωνοι με τη συνδίκη Λισαβόνα. Σα παρακαλώ και το λέω και στην έκθεσή μου να ακολουθήσετε τη λύση που προτείνω. Μεταβατική, ρεαλιστική, έστω προσωρινή, αλλά κυρίω Πρόεδρε δίκαιη. Σα ευχαριστώ όλου για τα ενδιαφέροντα που είπατε και για τη συνεργασία σα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Σιγητά. Εκείνη η συζήτηση ολοκληρώθηκε και η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 11.